Αγαπητοί συνάδελφοι, ε, χαίρομαι που σας βλέπω και ζητώ συγγνώμη για την κατανόησή σας. Ε, έπρεπε να συνεχιστεί το διαβημένο Προεδρείο να παρατεθεί η συνεδρίαση για πάρα πολύ ε, αναγκαστικούς λόγους και ανελημμένες υποχρεώσεις. Θέλω να ευχαριστήσω τον κύριο Συζήλμαση, Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο ε, που ενέκρινε αυτή την ε, αναβολή της συνεδρίασης στην καθυστερημένη έναρξη που δεν είναι και τόσο προφανές και αυτονόητο, ούτε ευχάριστο άλλωστε ε, και άκομψο από πλευρά μας που το κάναμε. Νομίζω ότι η Ένωση για τη Μεσόγειο θα αποκτήσει όλο και περισσότερη σημασία στις εργασίες της. Το έχουμε συζητήσει και στο παρελθόν πόσο σημαντικό είναι ε, και εμείς από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης να δώσουμε περισσότερη όθηση σε όλη αυτή την προσπάθεια. Και πιστεύω ότι και η σημερινή ε, απόφαση να προωθηθούν 29 έργα με 4 εκατομμύρια δισεκατομμύρια ευρώ είναι πάρα πολύ σημαντικό βήμα προς την κατεύθυνση αυτή. Και μετά την Υπουργική Διάσκεψη των χωρών της Νότιας Γειτονίας όπου συζητήθηκε και το θέμα αυτό τον Απρίλιο και το θέμα της γειτονίας έχουμε νέα δεδομένα. Στις 11 Ιουνίου εγκρίναμε την έκθεση Κούκαν στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο όπου και αποδίδουμε και μεγάλη σημασία στην περιφερειακή διάσταση της πολιτικής γειτονίας. Νομίζω ότι είναι εξαιρετική η σημασία αυτού και δεν το αμφισβητεί κανείς. Θα πρέπει να έχουμε διεθνή συνεργασία πέρα από σύνορα, πέρα από σύνορα και της Ευρωπαϊκής Ένωσης για να μπορούμε να έχουμε ειρηνική εξέλιξη και ειρηνική συνύπαρξη ε, και να μπορέσουν να προοδεύσουν και οι χώρες αυτές και κοινωνικά και οικονομικά. Και η κοινή μας αυτή οργάνωση, η Ένωση για τη Μεσόγειο, είναι το κατάλληλο μέσο και εργαλείο για να ε, επιτύχουμε την επιθυμητή πρόοδο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ που ήρθατε και σας παρακαλώ αμέσως να λάβετε το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι βουλευτέ, συνάδελφοι και φίλοι, χαίρομαι ιδιαίτερα που είμαι μαζί σας σήμερα για να σας παρουσιάσω, όπως είχε αποφασιστεί, την έκθεση πεπραγμένων της Γενικής Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο για το 2014 αυτό βέβαια είναι και μια ευκαιρία να μιλήσουμε και για την κατάσταση γενικότερα και την προοπτική της. Ε, χαίρομαι ιδιαίτερα διότι είχαμε δεσμευτεί κύριε Πρόεδρε με πολλούς ευρωβουλευτές στις συνεδριάσεις που κάναμε να παραμείνουμε σε μόνιμη επαφή με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ως Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο. Έτσι ώστε να μπορέσετε κι εσείς οι Ευρωβουλευτές μόνιμα να είστε πληροφορημένοι για τα αποτελέσματα των διαφόρων διαβουλεύσεων και εξελίξεων και θεμάτων που τίθενται ή προβλημάτων. Είναι για μένα σημαντικό θεσμικά, αλλά βέβαια και για το σύνολο της Ένωσης για τη Μεσόγειο να γίνει αυτή η αξιολόγηση, να πούμε πού βρισκόμαστε και βέβαια να δούμε τι θα κάνουμε και στο μέλλον. Σας προτείνω λοιπόν να γίνει μία παρουσίαση με μερικές διαφάνειες αλλά κυρίως ελπίζω να ακούσω ερωτήσεις σας για να μπορέσουμε έτσι να εμβαθύνουμε ορισμένες πτυχές του προγράμματός μας. Δεν ξέρω αν άρχισε η παρουσίαση, είναι εδώ στις δύο οθόνες. Καταρχήν θα ήθελα να σας υπενθυμίσω το θεσμικό πλαίσιο της Ένωσης για τη Μεσόγειο που είναι διακυβερνητική οργάνωση με 43 κράτη-μέλη και αυτό σημαίνει βέβαια δεν σημαίνει ότι περιοριζόμαστε στα διακυβερνητικά θέματα εξορισμού. Είμαστε ανοιχτοί σε εταιρικέ σχέσεις με το σύνολο των παραγόντων της περιοχής αυτής και με συγκεκριμένο στόχο την ενίσχυση, τη λειτουργική ενίσχυση της περιφερειακής συνεργασίας. Θα σας μιλήσω σήμερα βέβαια για την έκθεση πεπραγμένων της Γενικής Γραμματείας, αλλά θα ήθελα καταρχήν να τοποθετήσω την οργάνωση αυτή στο οικοσύστημά της που είναι πολύ πλούσιο γιατί δεν αφορά μόνο τα κοινοβούλια των χωρών μελών αλλά και άλλα θεσμικά όργανα. όπως το Αρλέμμα ή το Ίδρυμα Άννα Λίντ ή το Μίσνες Μέντα Ασκαμέ και τον ακαδημαϊκό τομέα. Δεν είναι εξαντλητική διαφάνεια, αλλά έχουμε ολόκληρο οικοσύστημα γύρω μας. Και θέλουμε να συνεργαστούμε περισσότερο και να συντονιστούμε με τους διάφορους άλλους θεσμούς που ενδιαφέρονται για τη ευρωμεσογειακή συνεργασία πώς διοικείται η Ένωση αυτή. Έχουμε κοινή ιδιοκτησία με την Συμπροεδρία που αποτελείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση για το Βορρά και χαιρετίζω εδώ ιδιαίτερα την παρουσία του φίλου μου Μαετρής Μακαμινή από την Υπηρεσία Εξωτερικών Τράσεων που εκπροσωπεί την Συμπροεδρία του Βορρά και φυσικά η Ιορδανία που είναι η νότια συμπροεδρία. Αυτή η έννοια της συμπροεδρίας είναι πολύ σημαντική γιατί έτσι μπορούμε θεσμικά πολιτικά να αναγνωρίσουμε ότι στα πλαίσια της Ευρωμεσογειακής Ένωσης χαράσεται ένα κοινό πρόγραμμα με κοινή ιδιοκτησία των προτάσεων και των λύσεων που αποφασίζονται από κοινού. Το σύνολο το διαχειρίζονται οι λεγόμενοι senior officials στην έδρα μας στη Βαρκελόνη. Θέλω όμως να τα πω και πιο συγκεκριμένα. Να δούμε ποιες είναι οι προκλήσεις και οι ευκαιρίες που διαθέτουμε στην περιοχή αυτή και τι προτάσεις κάνουμε για την εξέβρεση λύσεων και απαντήσεων. Νομίζω ότι στη διαφάνεια αυτή δεν χρειάζονται σχόλια διότι συνοψίζει ένα τμήμα των προκλήσεων που αντιμετωπίζουμε, όχι όλες βέβαια, οι κυριότερες ανεφαίνονται εδώ. Μερικές είναι πιο κεντρικές λοιπόν και θα ήθελα να τονίσω ιδιαίτερα το βασικό θέμα της απασχόλησης των νέων, ιδιαίτερα δε της ανεργίας αυτών που είναι κατεμένα κάτι πολύ ουσιώδες και ε, σημειώνεται κυριέτερα σε επίπεδο γυναικών. Έχουμε βέβαια προκλήσεις να αντιμετωπίζουμε αλλά και μέχρι το 2030 αντιμετωπίζουμε άλλες προκλήσεις. Πρέπει να σας πω βέβαια ότι οι προκλήσεις αυτές δεν περιορίζουν το όραμά μας. Το όραμά μας συμπεριλαμβάνει όχι μόνο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες που έχουμε για να υπάρξει εκεί μια εξισορρόπηση. Θα ήθελα λοιπόν να σας πω συνοπτικά ότι η εξέταση των προβλημάτων της, της κατάστασης της περιοχής πρέπει να συνδυάζει και τις προβλήματα και τις ευκαιρίες για να βρεθούν οι κατάλληλες απαντήσεις. Γι' αυτό να σας αναφέρω ποιες είναι οι δραστηριότητες της Γενικής Γραμματείας το γενικότερο της πλαίσιο σε σύγκριση με τις ευκαιρίες και τα προβλήματα αλλά και σε σύγκριση με την εντολή της. Η Γενική Γραμματεία έχει μια συγκεκριμένη εντολή η περιφερειακή συνεργασία να καταλήξει σε συγκεκριμένες και απτές δραστηριότητες με δύο άξονες. Πρώτον, τον διάλογο policy dialogue που λέμε και συγκεκριμένες προτάσεις με κοινωνικο-οικονομικές επιπτώσεις. Οι δύο αυτοί οι άξονες αποφέρουν τελικά αποτελέσματα ενθαρρυντικά και το λέω μετρημένα. Σε λίγο θα σας μιλήσω και για άλλα προβλήματα, αλλά τώρα θα ήθελα να σας πω ότι με τις δραστηριότητες του περιφερειακού διαλόγου Οργανώσαμε 8 υψηλού επίπεδου διασκέψεις, 13 συναντήσεις ανωτά των υπαλλήλων και πάνω από 100 συναντήσεις με εμπειρογνώμονες και στρογγυλές τράπεζες. με δικτύωση πάνω από 5.000 ενδιαφερομένων από, όλα τα επαγγελ... από όλους τους επαγγελματικούς ορίζοντες. Και όλα αυτά για να υπάρξει ένας καταλήτης που να καταλήγει σε συγκεκριμένα προγράμματα. Τα προγράμματα αυτά είναι 33 σήμερα. 33 σχέδια περιφερειακά. 50% από αυτά σήμερα έχουν αρχίσει ήδη να εφαρμόζονται θα συνεχίσουμε προφανώς να προσπαθούμε για την εφαρμογή και άλλων προγραμμάτων και σχεδίων. Βλέπετε εδώ την ε, γεωμετρική πρόοδο που έχει σημειωθεί, αλλά χρειάζεται ακόμη χρόνος και κάνουμε ό,τι μπορούμε ώστε η επίπτωση, η ορατότητα, τα αποτελέσματα να είναι όσο το δυνατόν σημαντικότερα και ουσιώδη για να συμβάλλουν στην επίλυση προβλημάτων ή για να εκμεταλλευτούμε τις υπάρχουσες δυνατότητες. Επίσης θα ήθελα να τονίσω ότι τα 33 αυτά σχέδια κατά περίπου 50% αυτό λίγο σχηματικά περίπου το 50% πραγματοποιούνται με δημόσιους οργανισμούς, κυβερνητικές υπηρεσίες ή διεθνείς οργανισμούς ή και χρηματοπιστωτικά ιδρύματα και 50% με μη κυβερνητικές οργανώσεις ε, της κοινωνίας των πολιτών, πανεπιστήμια, ιδιωτικό τομέα. Είναι πολύ σημαντικό να σημειώσουμε ότι υπάρχει τέτοιου είδους εξισορρόπηση. Επίσης η παρουσίαση αυτή μπορεί να διανεμηθεί αν θέλετε να την πάρετε ή όλοι για να έχετε τους αριθμούς μπροστά σας. 50% δημόσιο, 50% ιδιωτικό τομέα. Πολύ σημαντικό ώστε η Ένωση για τη Μεσόγειο να μπορέσει να συνεχίσει να λειτουργεί με όλους τους ενδιαφερόμενους της περιφέρειας και ιδιαίτερα με εκπροσώπους της κοινωνίας των πολιτών, ακαδημαϊκά δίκτυα, πανεπιστήμια κλπ. Οι δραστηριότητες, στα προγράμματα βασίζονται σε τρία κύρια θέματα, τα οποία θα αναφέρω σύντομα για να μην είναι υπερβολικά μακροσκελής η παρουσίαση. Πρώτη προτεραιότητά μας είναι η απασχόληση των νέων όπως είπα και πριν γιατί είναι ουσιώδες στοιχείο για την ανάπτυξη. Σε αυτή τη φάση τα διάφορα στοιχεία και δεδομένα για την προβληματική της ανεργίας ή απασχόλησης των νέων δεν χρειάζονται σχόλια. Πρέπει όμως να σημειώσουμε ότι η απασχόληση των νέων είναι θέμα σημαντικό και για τον νότο της Μεσογείου αλλά και για τον βορρά της και την Ευρωπαϊκή Ένωση στο σύνολό της. Και επομένω η απασχόληση των νέων είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό ώστε η Ευρώπη και ο Νότος της να μπορέσουν να συνεργαστούν Και το ιδεώδες βήμα για περιφερειακή συνεργασία είναι η δική μας οργάνωση με 13 προγράμματα μεταξύ των 33 που σας ανέφερα προηγουμένως, ειδικά για την απασχόληση των νέων και την ε, ανάπτυξη. Άλλη προτεραιότητα είναι οι γυναίκες. Ο ρόλος της γυναίκας στην κοινωνία και την κοινωνικο-οικονομική ζωή των χωρών του Νότου και εδώ αυτό ισχύει και για τον Νότο αλλά και για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Και το λέω γιατί βλέπω ότι γίνονται συζητήσεις πολλές φορές για το θέμα αυτό την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών στην κοινωνία. Εδώ έχουμε 10 προγράμματα ειδικά για αυτό το θέμα και από την Υπουργική Διάσκεψη του Παρισιού το 2013 μέχρι τώρα σημειώνεται μια πολύ σημαντική δυναμική και δραστηριότητες με βάση τη Βαρκελόνη με πολλούς ενδιαφερόμενους multi-stakeholder ώστε τα 10 αυτά προγράμματα να στοχεύσουν 50.000 ανθρώπους που ήδη εφαρμόζουν αυτά τα προγράμματα. Τρίτη προτεραιότητα, η βιώσιμη ανάπτυξη, η οποία κυρίε και κύριοι πρέπει να τη δείτε ευρέως. Δηλαδή ενέργεια, κλιματολογικές αλλαγές, περιβάλλον, είδωρ. Η βιώσιμη ανάπτυξη ευρύτατα θεωρούμενη δηλαδή και εδώ συνεργασία και περιφερειακό διάλογο προωθούμε στα προγράμματα μας. 14 τέτοια προγράμματα υπάρχουν για το θέμα αυτό της βιώσιμης ανάπτυξης που μας επιτρέπουν να το αντιμετωπίσουμε. Ιδιαίτερα θα ήθελα να τονίσω την βιώσιμη αστική ανάπτυξη, ανάπτυξη των πόλεων και νομίζω ότι το θέμα αυτό θα ε, συναντήσει όλο και περισσότερη, θα έχει όλο και περισσότερη σημασία στο μέλλον. Αυτά τα κάνουμε με βάση ένα δίκτυο. Η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι διακυβερνητική οργάνωση σας είπα, αλλά δεν μπορούμε ούτε πρέπει να εργαζόμαστε, να λειτουργούμε μόνοι μας σε απομόνωση αφού ο κύριος στόχος μας είναι η δημιουργία συνεργειών και συνεργασίας. Χαιρετίζω εδώ τις σχέσεις που έχουμε δημιουργήσει με τα κοινοβούλια, δηλαδή την Κοινοβουλευτική Συνέλευση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, που οργάνωσε τρεις διασκέψεις στη Βαρκελόνη, στο, στην έδρα δηλαδή, με την Πολιτική, Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και επίσης μια πολύ καλή διάσκεψη ολομέλειας στη Λισαβόνα πριν από λίγες εβδομάδες με διάσκεψη των Προέδρων που ήταν πολύ μεγάλη επιτυχία. Επίσης συνεργαζόμαστε με χρηματοπιστωτικά ιδρύματα διεθνή και με την κοινωνία των πολιτών, πανεπιστήμια και άλλους ώστε να είναι ως το δυνατόν ευρύτερη η προσέγγιση και να συνδέει το top-down με το bottom-up ώστε να έχουμε και στρατηγική άποψη χωρίς να ξεχνάμε την καθαρά πολιτική. Δηλαδή η στρατηγική αντιμετώπιση να είναι λειτουργική και πραγματιστική, ρεαλιστική και ευρύτερη. Θα καταλήξω τώρα την παρουσίασή μου λέγοντας ότι πέρα από την έκθεση πεπραγμένων του 14 δεν θα μπορούσα να είμαι πολίτης της Μεσογείου, είμαι Μαροκινός, είμαι από το Μαχρέμπ, είμαι Μεσογειακός. Τρία, τρεις ιδιότητες με τις οποίες δεν μπορώ να σας πω ότι αρκούν αυτά που κάναμε. Θα ήθελα να σας πω πόσο σημαντικό είναι να δούμε το μέλλον βλέποντας όχι μόνο που βρισκόμαστε, αλλά και το σύνολο των προκλήσεων, των προβλημάτων που αντιμετωπίζουμε. Και σε αυτόν τον δρόμο του μέλλοντος θα ήθελα να κάνω τις εξής προτάσεις. Πρώτον, το και βασικότερον, τώρα που γιορτάζουμε την 20η επέτειο της διακασίας της Βαρκελόνης, Το Νοέμβριο δηλαδή θα συμπληρωθούν, όπου το χρονοδιάγραμμα εργασιών της Ευρώπης προβλέπει την αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας για το φθινόπωρο, τη στιγμή όπου και ο ΙΕ επανεξετάζει τους στόχους της χιλιετίας, σε λίγες εβδομάδες, τη στιγμή όπου συμπίπτουν όλα αυτά τα χρονοδιαγράμματα θα ήθελα εδώ να τονίσω την ανάγκη που υπάρχει να ξανατονίσουμε τη σημασία της περιφερειακής διάστασης της συνεργασίας. Η περιφερειακή διάσταση που παραμένει αδύναμος κρίκος, διότι όλες οι μελέτες δείχνουν ότι δεν αρκεί ο βαθμός περιφερειακής συνεργασίας που υπάρχει, ενώ η λύση είναι προφανής. Να συνεργαστούν όλες αυτές οι χώρες και οι χώρες του Νότου μεταξύ τους αλλά και οι χώρες του Νότου με τις βόρειες χώρες με την Ευρωπαϊκή Ένωση ώστε να υπάρξει πραγματικό region building. Είναι κάτι ιδιαίτερα σημαντικό να μην το ξεχνάμε και να ενδυναμώνουμε την περιφερειακή διάσταση που μας φαίνεται βασικότατο θέμα. Επίσης σημαντικό είναι μαζί από κοινού να ενδυναμώσουμε την ορατότητα τά των δράσεών μας για να υπάρξει όπως λέμε κοινή ιδιοκτησία των αποτελεσμάτων και να ακούσουμε όλα τα συνεργαζόμενα ιδρύματα και από πλευράς Γενικής Γραμματείας της Ένωσης για τη Μεσόγειο ιδιαίτερα θεωρούμε ότι η κοινή εργασία, η συνεργασία μαζί σας κύριοι βουλευτέ είναι πολύ σημαντική με ένα όραμα που επιβεβαιώνει τις επιλογές που ήδη έχουμε κάνει, δηλαδή την απασχόληση των νέων, τη βιώσιμη ανάπτυξη και την ενδυνάμωση του ρόλου των γυναικών, αλλά με επιτάχυνση της κίνησης αυτής. Σήμερα γίνεται. Έχουμε 33 προγράμματα και σας διαβεβαιώνω ότι μπορούμε εύκολα να διπλασιάσουμε και να τριπλασιάσουμε τον αριθμό αυτών. Αλλά γι' αυτό χρειάζεται περισσότερη πολιτική στήριξη, οικονομική στήριξη και μεγαλύτερος συντονισμός και συνεργασία μεταξύ των διαφόρων παραγόντων της συνεργασίας ώστε να μπορέσουμε να προχωρήσουμε μαζί. Καταλήγω αναφέροντας τρία, τρεις προτάσεις που νομίζω ότι είναι πολύ σημαντικές. Όταν θα επανέλθω ίσως την επόμενη χρονιά για την έκθεση δραστηριοτήτων του 2015 θα σας μεταφέρω τα πρώτα αποτελέσματα για τις δράσεις τις οποίες προτείνουμε. Καταρχάς θα πρέπει να ξεκινήσουμε μια μεγάλη πρωτοβουλία πάνω στα θέματα της ανάπτυξης και της μετανάστευσης. Νομίζω ότι το θέμα της μετανάστευσης που είναι το μεγάλο θέμα σε αυτή τη φάση δεν μπορεί να ειδωθεί αποκλειστικά σε επίπεδο δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Απαιτείται να το δούμε ευρύτερα, μακροπρόθεσμα, να εντάξουμε τη διάταξη της ανάπτυξης. Τότε μόνο θα μπορέσουμε κάτι να πετύχουμε. Και δεν υπάρχει καλύτερος χώρος από την Ένωση για τη Μεσόγειο για να ξεκινήσει μια τέτοια πρωτοβουλία σε συνεργασία με άλλους. Το λέγω αυτό, είναι κάτι το οποίο βέβαια θα το θέσω σαν πρόταση στην διάσκεψη των Προέδρων, διότι αυτοί είναι που θα πρέπει να πάρουν τις απαιτούμενες αποφάσεις. Πιστεύω επίσης ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο. Πέρα από τα λόγια, οι άνθρωποι, οι πολίτες, οι πληθυσμοί θα πρέπει να κατανοούν ο ένας τον άλλο καλύτερα. Δεν θα πρέπει εμείς να δεχθούμε να υπάρχει ένα ρήγμα πολιτισμικό, μια διαταραγμένη πολιτιστική επικοινωνία. Πρέπει να επιμείνουμε λοιπόν εδώ και η πρωτοβουλία του Ισπανού Επουργού Εξωτερικών Υποθέσεων είναι καλή τον Ιανουάριο ξεκίνησε οργανώνοντας στην Βαρκελόνη, στην έδρα της Ένωσης για τη Μεσόγειο, μια μεγάλη συνεδρίαση για τον διαθρησκευτικό διάλογο. Κλείνοντας, θα ήθελα να πω ότι θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο σε ετήσιες συναντήσεις όλων των οργανώσεων που κινητοποιούνται στη Μεσόγειο για να μπορέσουμε να συντονίσουμε καλύτερα τις προσπάθειές μας να αναπτύξουμε τις συνεργίες μας και, τις, και να αποφύγουμε επικαλύψεις. Αυτά θα ήθελα να σας πω. Επιτρέψτε μου συμπερασματικά να με κάπως ουμοριστικό τρόπο είδα αυτή την γελιογραφία στη Herald Tribune βλέπουμε κάποιον ο οποίος είναι έτοιμος να ανατιναχθεί, να αυτοκτονήσει και ο οποίος βλέποντας όμως ότι υπάρχει μια ταμπέλα στο μαγαζί που λέει ότι υπάρχει δυνατότητα πρόσληψης υπαλλήλων, ζητούνται υπάλληλοι, ε, λέει αχ ευτυχώς που θα μπορέσω να δουλέψω και έτσι δεν θα την αυτό στον αέρα. Euh, Ευχαριστώ πολύ κύριε Γενική Γραμματέα. Ε, ε, κύριε εσείς σας συγχαίρω, έχετε συμπληρώσει τριετία στην ε, Βαρκελόνη, αναφερθήκατε στις προτεραιότητες και η απασχόληση είναι μία από αυτές. Επίσης η ενδυνάμωση και χειραφέτηση των γυναικών, μεγαλύτερος ρόλος τους στην κοινωνία, βιώσιμη ανάπτυξη είναι η τρίτη. Βλέπω ότι ενδιαφέρονται πολλοί συνάδελφοι όπως και εγώ και θέλουμε περισσότερες λεπτομέρειες να μάθουν πώς μπορεί η Ένωση για τη Μεσόγειο να καταπονεμήσει την ε, λάθρο μετανάστευση και εσείς ε, από το Μαρόκο όπου ε, προσφάτως έχει καταστεί χώρα ε, όχι μόνο ε, διέλευσης αλλά και προορισμού. Θα ε, δούμε λοιπόν την συνεργασία και μετά τη Λισαβόνα κτλ. Λοιπόν, αγαπητοί συνάδελφοι, νομίζω θα πρέπει να ορίσουμε ένα δίλεπτο χρόνο αγόρευσης γιατί έχουμε ήδη καθυστερήσει. Θα δώσω πρώτα το λόγο στο συνάδελφο Μιγιάν Μον. Ευχαριστώ Πρόεδρε, ευχαριστώ και το Γενικό Γραμματέα της Ένωσης για τη Μεσόγειο που ήρθε για άλλη μια φορά εδώ, νομίζω και πέρυσι. Πριν από 14-15 μήνες είχαμε τη τύχη να τον υποδεχθούμε εδώ και το ξαναβλέπουμε σήμερα. Τον ευχαριστώ ε, για το ενδιαφέρον που δείχνει να έχει διάλογο με την Επιτροπή μας και με το Κοινοβούλιο. Θέλω επίσης να τον συγχαρώ, διότι όταν το περιφερειακό πλαίσιο είναι τόσο δύσκολο και το πολιτικό και το οικονομικό, ε, λόγω και της πρόσφατης κρίσης που έπληξε και ε, τους προϋπολογισμούς πολλών κρατών αλλά και πολλών διεθνών οργανισμών είναι 36, 33 συγγνώμη, τα έργα που τρέχουν και γύρω στα 50 που ολοκληρώνονται. Πραγματικά είναι αξιέπαινη αυτή η εκτέλεση των έργων που είναι από ε, τις βασικές εντολές της Γενικής Γραμματείας. Μας μιλήσατε για μια χρονική σύμπτωση φέτος. Ναι, είναι γεγονός αυτό. Είναι παρόν ο Έντουαρτ Κούκαν, συγητή τη έκθεση για την πολιτική γειτονία, ακριβώ εδώ στο Κοινοβούλιο και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αλλά και η Υπηρεσία Εξωτερική Δράση. Ε, μελετούμε αυτόν τον καιρό την ανανέωση της πολιτικής γειτονίας και θα ήθελα να ακούσω από τη δική σας προνομιούχα θέση όπου έχετε την ευκαιρία να παρακολουθείτε εκ του σύνεγης ε, αυτή τη γειτονία. Τι θα μας ε, προτείνατε, τι αλλαγές χρειάζονται, καινοτομίε, μεταρρυθμίσεις, μετασχηματισμοί, τι πρέπει να αλλάξει στην πολιτική γειτονία ε, που εξετάζει και μελετά η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης και το Κοινοβούλιο θα αποφανθεί σε λίγες εβδομάδες. Ευχαριστώ η κυρία Γκόμες για δύο λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ κύριε Γενική Γραμματεύ για την παρουσίασή σας. Συμφωνώ απολύτως με τις προτεραιότητες που έχετε θέσει. Το θέμα της εργασίας των νέων είναι κομβική σημασία και για το βορρά και για το νότο της Μεσογείου. Ε, βεβαίως οι εξουσίες στις γυναίκες και η χειραφέτησή τους, το empowerment όπως λέγεται στα αγγλικά, και σας συγχαίρω γι' αυτό, ίσως θα πρέπει να επενδύσουμε περισσότερο στην κοινοβουλευτική διάσταση. Παράδειγμα, να εμβαθύνουμε τον διαπολιτισμικό και διαθρησκευτικό διάλογο σε κοινοβουλευτική βάση. Νομίζω θα ήταν πολύ χρήσιμο να έχουμε κοινά σχέδια και έργα. Οι βουλευτές, επαναλαμβάνω, από τις δύο όχθες της Μεσογείου ας πούμε με επισκέψεις σε συγκεκριμένα έργα ή πρωτοβουλίες διαλόγου για να γνωριστούμε καλύτερα, να εμβαθύνουμε σε ένα διάλογο που κάνουμε ήδη σε επίπεδο κοινοβουλευτικής συνέλευσης, αλλά ε, έχει φανεί και ότι υπάρχει και περισσότερο έδαφος για εμβάθυνση. Λοιπόν, θα ήθελα να σας ρωτήσω το εξή ε, γίνεται λόγος για τη μετανάστευση και για τη λεγόμενη παράτυπη μετανάστευση. Τίποτα δεν αφήνει να εννοηθεί ότι θα βελτιωθεί η κατάσταση. Το αντίθετο μάλιστα. Γιατί έχει να κάνει και με όλες τις σειράξεις αυτό που σοβούν ε, ε, στη γειτονιά μας, αλλά και παραπέρα. Εσείς πιστεύετε ότι το γεγονός ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν συζητάει τον νόμιμο τρόπο να φτάνουν οι μετανάστες Πώς το βλέπετε, μήπως αυτό θα ήταν ένας τρόπος να χαλιναγωγηθούν ε, αυτά τα φαινόμενα παράτυπης μετανάστευσης με όλα τα συμπαραμαρτούντα και τις ε, πτυχές ασφάλειας. Σε ό,τι αφορά λοιπόν την περιφερειακή διάσταση, την οποία επίσης αναφέρατε, τι θα μπορούσαμε να κάνουμε για να επενδύσουμε στη σχέση νότου-νότου. Ας πούμε Αλγερία-Μαρόκο. Εάν ε, ε, συνεργάζονταν δύο χώρε αυτές θα μπορούσε να είναι τεράστια διαφορά. Ευχαριστώ. Ο κύριος Αουστριβίτσιο, παρακαλώ. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Θέλω να συγχαρώ τον Γενικό Γραμματέα για την παρουσίασή του και για την επιθυμία του να συζητήσει τα θέματα αυτά μαζί μας. Είναι καλό να ανταλλάσσουμε τις εμπειρίες μας και να βλέπουμε πως έχουν τα διάφορα θέματα όπως τα βλέπουν τα περιφερειακά όργανα. Έχουν προχωρήσει σε συγκεκριμένα πρακτικά προγράμματα και αυτό είναι πολύ σημαντικό. Αυτό θέλει ο καθημερινός πολίτης, ο απλός πολίτης να βιώσει. Έχω δύο ερωτήσεις. τις οποίες ίσως να μπορέσετε να είσαστε πιο αναλυτικός. Για τα θέματα της πολιτικής συνεργασίας μιλήσατε για την κοινοβουλευτική συνέλευση της Ένωσης. Είπατε για τις τακτικές συναντήσεις τις οποίες οργανώνει η συνέλευση αυτή. Σε ποιο βαθμό η συνέλευση αυτή, η σύνθεσή της, η ολομέλειά της, οι επιτροπές της αντικατοπτρίζουν την πραγματικότητα. Υπάρχει δυνατότητα να καταστεί πιο αντιπροσωπευτική μέσω περαιτέρω δραστηριοτήτων. Μπορεί σε κοινοβουλευτικό επίπεδο να ενισχύσει την περιφερειακή συνεργασία με μια νέα όθηση. Και δεύτερον το λεγόμενο αίσθημα του ανήκειν. Σε ποιο βαθμό οι εμπλεκόμενες χώρες, ιδιαίτερα οι χώρες της νότιας πλευράς της Μεσογειακής Λεκάνης, αισθάνονται ότι πράγματι εμπλέκονται, ότι πράγματι είναι ιδιοκτήτες αυτής της Ένωσης. Έχει μεγάλη σημασία να μην επιβάλλει κανείς μια τέτοια εταιρική σχέση, αλλά να συμφωνεί και να εφαρμόζει τα θέματα αυτά σε επίπεδο συνεργασίας. Θέλω να μας μιλήσετε λοιπόν για την αίσθηση που έχουν οι χώρες μέλη. Ο Καστάλντο έχει ζητήσει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θα ήθελα και εγώ να καλωσορίσω τον αξιότιμο Γενικό Γραμματέα. Μεγάλη χαρά για μας να σας συναντούμε ξανά και να μπορέσουμε να ανταλλάσσουμε απόψεις. Κατανοείτε βέβαια ότι συμφωνώ με τις προτεραιότητές σας, ιδιαίτερα για αυτά τα οποία είπατε για τον διαθρησκιακό διάλογο και τον διαπολιτισμικό διάλογο και για τον τρόπο με τον οποίο θα ασχοληθούμε με το κεντρικό θέμα σήμερα, το θέμα δηλαδή της μετανάστευσης. Είπατε ότι θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πρόβλημα αυτό με σφαιρικότερο τρόπο και όχι αποκλειστικά σε θέμα δημόσιας τάξης και ασφάλειας. Η άμεσή μου λοιπόν θα είναι ο λίγων ξερή και άμεση. Ξέρετε ότι η αποστολή Εουμπαφορμέντ εγκρίθη από το Συμβούλιο. Αν θυμάμαι καλά, είχε πέντε σκάφη στη διάθεσή της και διάφορα άλλα μέσα και είχε μια συγκεκριμένη εντολή. Σήμερα επίσης υπήρξαν στη Μεσόγειο ένας νεκρός και ένας τραυματίας σε ένα σκάφος που ξεκίνησε από τη Λιβύη και δεν ξέρουμε ποιος είναι υπεύθυνο για αυτό το συμβάν. Η εισαγγελία του Ακράγαντα στη Σικελία ξεκίνησε μια έρευνα για πιθανότητα δολοφονίας. Και νομίζω ότι το ερώτημα το οποίο τίθεται είναι το εξής. Θεωρείτε εσείς ότι η συγκεκριμένη αποστολή στα πλαίσια της εντολής που έχει δοθεί από το Συμβούλιο είναι κατάλληλη και ανταποκρίνεται στις προτεραιότητές σας. Βρίσκεται στο ύψος των προτεραιοτήτων σας. Ή πρέπει να υπάρξουν περαιτέρω βελτιώσεις και κριτικές. Σας εύχομαι καλή προσπάθεια. Ο κύριος Κουκάν έχει το λόγο. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Ζητώ συγγνώμη για την καθυστέρηση. Θα ήθελα να καλωσορίσω το Γενικό Γραμματέα από πλευρά μου και εγώ. Τους τελευταίους μήνες είναι πιο συχνός επισκέπτης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μας χαροποιεί αυτό όλο και περισσότερο συζητούμε μαζί του, όλο και περισσότερο, τόσο περισσότερο έχουμε την ευκαιρία να εκτιμούμε το δικό του έργο και της Γενικής Γραμματείας συνολικότερα. Ναι. Πολύ σύντομα θα ήθελα να φέρω ότι η Επιτροπή μας ήδη έχει ψηφίσει την έκθεση για την αναθεώρηση πολιτικής γειτονίας η Ένωση για τη Μεσόγειο και η Γενική Γραμματεία αναφέρεται στην έκθεση αυτή, γι' αυτό είμαστε πολύ ευγνώμονες για όλα τα συγκεκριμένα στοιχεία που μας παρουσιάσατε σήμερα, τα ενημερωτικά. Πραγματικά εκτιμούμε ότι ασχολείστε με συγκεκριμένο έργο ε, δεδομένου του χαρακτήρα της οργάνωσης και της σύνθεσης ε, και των μελών δηλαδή. Θέλω να πω όμως ότι η έκθεση αυτή μπορεί να χρησιμοποιηθεί για ένα πλαίσιο για τη μελλοντική συνεργασία ε, και να συνδεθεί η Ανατολική με την Νότια γειτονία και να επικεντρωθούμε στα πολύ συγκεκριμένα χειροπιαστά έργα. Εμένα δεν μου αρέσουν τα μεγαλόστομα λόγια, οι δηλώσει κτλ. Οποιοδήποτε συγκεκριμένο έργο μπορεί να χρησιμοποιηθεί, να εκτελεστεί, είναι πρόσδεκτο και θα βοηθήσει. γιατί εκεί έχουμε συγκεκριμένα αποτελέσματα και αυτή τη στιγμή ολοκληρώνονται τα μικρά έργα, μπορούν να ακολουθήσουν και τα μεγαλύτερα. Σας ευχαριστώ που ήρθατε και πάλι και προσβλέπω στη συζήτηση για τη συνεργασία ε, των δύο οργανισμών μας. Ευχαριστώ, Έτβαρτ. Ο συνάδελφος τον Ίνο Πίτσουλα, παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ. Κύριε Γενική Γραμματέως, πρώην μέλος της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης της Μεσογείου, βλέπω ότι ασχολείστε με τα θέματα αυτά, μετανάστευση, δημογραφική αλλαγή, εκπαίδευση, παιδεία, χρηματοδότηση μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ισότητα φύλου και πιο σημαντικό δεν είναι μόνο η απασχόληση, αλλά ε, το να δοθεί ε, η δυνατότητα ουσιαστικής παρέμβασης των νέων και αυτό είναι παράγον σταθερότητας. Γίνονται κλήσεις για να δημιουργηθεί μια ζώνη ελευθέρων συναλλαγών στη Μεσόγειο και να ενισχυθεί η συνεργασία και οι εμπορικές συναλλαγές των χωρών του Νότου μεταξύ τους. Ε, τι άποψη έχετε γι' αυτά. Και ε, τι γίνεται με τις επενδύσεις στις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Χρειάζεται συνεργασία ε, με την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης και άλλα διεθνή μεγάλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Ευχαριστώ κύριε Πίτσουλα. Η κυρία Ευχαριστώ πολύ κύριε Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Γενικέ Γραμματεύ, με μεγάλη χαρά σας άκουσα και είδα την παρουσίασή σας που είναι πολύ θετική. Θέλω όμως να σας πω κάτι που το γνωρίζετε. Οι προκλήσεις που πρέπει να αντιμετωπίσουμε σήμερα στη Μεσόγειο είναι τεράστιες. Το θέμα των σειράξεων, των πολέμων, του φανατισμού της μετανάστευσης, της ασφάλειας, της σταθερότητας για ορισμένες χώρες. Όλα αυτά είναι τεράστιες προκλήσεις και νομίζω ότι φυσικά είναι θετική η έκθεσή σας, αλλά δεν ζούμε σε κανονικούς καιρούς σήμερα. Και γι' αυτό αναρωτιέμαι μήπως δεν θα έπρεπε να σκεφτούμε την αλλαγή, την εξέλιξη της εντολής που χρειάζεται η Ένωση για τη Μεσόγειο ώστε με, όλους τους, ε, με όλους τα θεσμικά όργανα της Ένωσης να προσπαθήσει να λύσει σε κάποιο βαθμό όλα σε αυτές τις προκλήσεις. Και έπειτα έχω και δύο σύντομα ερωτήματα. <clears throat> Το πρώτο. Θεωρείτε ότι η απουσία μεταναστευτικής πολιτικής για την Ευρώπη ή όση πολιτική υπάρχει είναι σωστή και δεύτερον η πολιτική ανάπτυξης που έχουμε εφαρμόσει έχει αποφέρει καρπούς ή πρέπει να αναθεωρηθεί. Ξέρω ότι δεν θα τα λύσουμε όλα διαμίας, αλλά πρέπει νομίζω να επανεπικεντρωθούμε σε αυτά τα θέματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κυρία κύριος Μπεργαμίνη τελευταίος. Ορίστε. Από την Υπηρεσία Εξωτερικών Δράσεων για τη Μεσόγειο. Είμαι σύντομος. Θα ευχαριστήσω το Γενικό Γραμματέα, τον κύριο Σιζιλ Μάτσι. Συνεργαζόμαστε και με την Ιορδανική Προεδρία εδώ και τρία χρόνια και τέσσερις μήνες Θέλω να υπογραμμίσω εδώ σε ποιο βαθμό η Ένωση για τη Μεσόγειο είναι κάτι το μοναδικό, ένα μοναδικό φόρουμ. Και όχι μόνο μοναδικό, αλλά και απαραίτητο. Ε, είναι το πυρήνας της προσπάθειάς μας είναι ο αγώνας για τους νέους, ο αγώνας για την απασχόληση ανάμεσα σε τόσες πολλές χώρες, 43 χώρες. Ελπίζουμε λοιπόν ότι ίσως σε κάποια φάση θα μπορέσουμε να αναθεωρήσουμε τις μεθόδους εργασίας μας, αφού προσμετρήσουμε τις προσπάθειες που έγιναν τα τελευταία τρία χρόνια σε πολιτικό επίπεδο. Θα σας δώσω συνοπτικά δέκα λόγους για τα πλεονεκτήματα της Ένωσης και για τις ανάγκες στήριξης από τις 43 πρωτεύουσες. Πρώτον, είναι το μοναδικό φόρουμ όπου η Παλαιστίνη με το όνομα Παλαιστίνη έχει έδρα και συνεργάζεται με το κράτος του Ισραήλ. Δεύτερον, έχουμε σε επίπεδο υψηλών στελεχών υπαλλήλων, σε καθημερινό επίπεδο αλλά και σε επίπεδο πρέσβεων σε δίμενη βάση, εκπροσώπους της Άγκυρας, της Τουρκίας και της Κύπρου που συνεργάζονται επίσης ε, με αυτά τα οποία είπα. Φυσικά και της Ελλάδας. Ταυτόχρονα η κυβέρνηση της, Αλε... της ε, Αλγερίας συνεισφέρει οικονομικά στην λειτουργία της Γενικής Γραμματείας ε, η οποία διοικείται γραμματεία από έναν μαροκινό διπλωμάτη, θαύμα διπλωματικό δηλαδή, για τη Λιβύη. Είχαμε οργανώσει εδώ και αρκετό καιρό μια συνάντηση και είχαμε τον Ισραηλινό Υπουργό Μεταφορών και τον Λίβιο Υπουργό Μεταφορών. Για πρώτη φορά από το 1948 υπήρξε μια τέτοια μορφή επικοινωνίας. Για την Συρία είναι μία από τις λίγες κοινέ θέσεις τις οποίες καταλήγουν τα κράτη-μέλη λέγοντας ότι δεν θα πρέπει εμείς να αφήσουμε την έδρα της Συρίας χειρεύουσα όχι βέβαια τη Συρία του Μπασάρ Ελασάντ, αλλά ούτε καν ακόμη τουλάχιστον την Συρία της αντιπολίτευσης. Ε, για τις γυναίκες, ε, ο κύριος της Ζηλμασής σας μίλησε για το ρόλο των γυναικών ήδη από το 1993, συγγνώμη 2013 τέθηκε το θέμα, σε συνεργασία με ορισμένες αραβικές πρωτεύουσες τις οποίες υπάρχουν συντηρητικές μουσουλμανικές ηγεσίες Μέχρι τώρα αυτά τα υπουργικά συμπεράσματα παραμένουν ιδιαίτερα φιλόδοξα σε επίπεδο δικαιωμάτων γυναικών, θέσεις γυναικών στην οικονομία και καταπολέμησης της βίας. Οι χώρες του Ευρωπαϊκού Νότου για πρώτη φορά ε, φιλοξενούν συναντήσεις της Ένωσης, η Λιθουανία πριν ε, ένα χρόνο και θα τελειώσω τώρα με δύο επιπλέον σημεία. Χάρη στην Ένωση για τη Μεσόγειο, σε επίπεδο πολιτικής ολοκλήρωσης, οι ευρωπαϊκές χώρες συμφώνησαν να πάνε πιο πέρα από τη συνθήκη της Λισαβόνας. Έχουμε συνεδριάσεις υπουργών όπου προεδρεύουν περιφερειακοί επίτροποι. Και τέλος, όπως είπε ο κύριος Γενικός Γραμματέας, προσπαθούμε εμείς να δημιουργήσουμε την αίσθηση της συνδιεύθυνσης και της συνδιαχείρισης με το βασίλειο της Ιορδανίας. Αυτή η διπλή δικέφαλη αν θέλετε μορφή διοίκησης εκφράζεται πλήρως και εδώ συμφωνώ με τον Ιουσέφ Μπαταϊνέ και εκφράζω και τις απόψεις του, τον πρέσβη της Ιορδανίας. Και νομίζω ότι η κατάσταση αυτή μπορεί να οδηγήσει στην αναθεώρηση της πολιτικής γειτονίας. Βρίσκεται στην καρδιά της απασχόλησής μας σήμερα το θέμα της Μεσογείου. και οι χώρες της Μεσογείου εν πολλής καταλήγουν σε κοινά συμπεράσματα και σε σχέση με την καταπολέμηση της τρομοκρατίας, ειδική στην προστασία του περιβάλλοντος, ειδική στην επιχειρηματικότητα, ειδική στον ακαδημαϊκό πανεπιστημιακό χώρο. Η προτεραιότητα πρέπει να δοθεί στους πολιτικούς. Θα δώσω το λόγο στην κυρία Λιωμάθη σύντομα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Πολύ γρήγορα. Επειδή έχω συμμετάσχει στις συζητήσεις που κατέληξαν στην ίδρυση της Ένωσης για τη Μεσόγειο, θα ήθελα μόνο να θυμίσω το εξής. Η ιδέα αυτή προέκυψε και από μία διαπίστωση ότι η Ευρώπη ακόμα και αν θέλει να έχει ένα ειδικό βάρος οικονομικό και πολιτικό στον αυριανό κόσμο, δεν έχει την απαραίτητη ε, ούτε οικονομική ούτε γεωγραφική διάσταση από μόνη της. Οπότε, ε, κατέρωθεν της Μεσογείου ε, και οι δύο πλευρές δεν έχουμε απλώς την επιθυμία αλλά και την ανάγκη να ενωθούμε για να έχουμε μεγαλύτερο ειδικό βάρος παγκοσμίως για να φτάσουμε στα 700 εκατομμύρια κατοίκους που είναι μια κρίσιμη μάζα για να αντιμετωπίσουμε ε, την, ε, τον ανταγωνισμό ή την ηγεσία άλλων μεγάλων ε, σχηματισμών παγκοσμίω. Δεν θα πρέπει ποτέ να το λησμονούμε αυτό και είναι κοινό μας στόχος και να μην το ξεχνάμε ποτέ. Θα πρέπει να είμαστε αρκετά ομοιογενείς και να έχουμε αρκετά ισχυρούς δεσμούς για να μπορούμε να βαρύνουμε ως δύναμη ευρωμεσογειακή δύναμη παγκοσμίω. Αυτό έχει σημασία. Κύριε Γενική Γραμματέα, βέβαια, το ζήτημα αυτό είναι άκρος πολιτικό. Δηλαδή, είστε το εξή ερώτημα. Μήπως έχουμε οδηγηθεί σε μια πολιτική αποτελμάτωση. Βεβαίως έχω σημειώσει πολύ προσεκτικά όλα αυτά που κάνατε και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά υπάρχει ένα πρόβλημα. Δεδομένων των σειράξεων που έχουμε γύρω από τη Μεσόγειο, ε, έχουμε την εντύπωση ότι αυτό το ιδεώδες και αυτή η βούληση κάπως υποχωρούν ε, σε σχέση με το πλαίσιο της λήψης αποφάσεων που πριτάνευσε όταν ιδρύθηκε η Ένωση για τη Μεσόγειο, που πιστεύω ότι είναι από τις ε, πιο σπουδαίες ιδέες για τον αυριανό κόσμο. Ευχαριστώ κύριε Υπουργέ. Παρακαλώ κύριε Γενικέ Γραμματεύ για να κλείσετε. 5-7 λεπτά. Για όλη τη Μεσόγειο 5 με 7 λεπτά. Καλά θα ξανάρθετε, δεν θα τα πείτε όλα τώρα. Ευχαριστώ. Κύριε και κύριοι, σας ευχαριστώ για τα ενθαρρυντικά σας λόγια, διότι ενδιαφέρον μόνο άκουσα υποστήριξη, ενθάρρυνση, βούληση, επιθυμία. Δεν σημαίνει αυτό καθόλου όμως συγκατάβαση, ε, ούτε επιταγή ε, λευκό για ό,τι κάνουμε. Ε, πάντως όλα αυτά που άκουσα τα θεωρώ ενθάρρυνση και έντονο ενδιαφέρον για την περιοχή και την περιφέρειά μας. Είναι πάρα πολύ σημαντικό για μας να σας ακούμε να λέτε όλα αυτά που είπατε και όλα που ακούσαμε και σας διαβεβαιώ ότι τα σημείωσα πάρα πολύ προσεκτικά. Ε, δεύτερον, έχω επίγνωση της πολυπλοκότητας του γενικότερου περιβάλλοντος και πλαισίου, αλλά σήμερα ήρθα εδώ να σας πω ότι η Μεσόγειος έχει διεύθυνση και τηλέφωνο και mail και μπορείτε να απευθυνθείτε σε Αυτό δεν σημαίνει ότι έχουμε ένα μαγικό ραβδί για να τα λύσουμε όλα. Αυτό θα ήταν πάρα πολύ ωραίο και θα ήταν και πάρα πολύ ε, υπερφύαλο από πλευρά μα να το ισχυριστούμε. Αλλά στην ευρωμεσογειακή συνεργασία στο παρελθόν έλειπε αυτό το μέσο, αυτό το εργαλείο για να παρακολουθεί, να πλαισιώνει και να ε, ενεργεί. Και για μένα είναι σημαντικό αυτό. Θέλω να συνεργαστούμε για να συνεχίσουμε να κινητοποιούμε την ομάδα αυτή που εδρεύει στη Βαρκελόνη και απαρτίζεται από 60 μέλη και θέλω να σας αποτίσω ένα φόρο τιμής διότι είναι αφοσιωμένοι, αποτελεσματικοί, ε, αξιόλογοι και θέλω ε, ενώπιόν σας να εξαρώ αυτή τους τη συνεισφορά. φαντάζομαι και εγώ ότι θα ρωτούσατε πολλά για τη μετανάστευση, οπότε έχω προετοιμαστεί κιόλας να απαντήσω, αλλά Εκτός αυτού, θα ήθελα να σας μιλήσω όχι μόνο ως Γενικός Γραμματέας, αλλά και ως πολίτης από τη Μεσόγειο. Δεν σας ομιλεί εδώ ο Μαροκινός διπλωμάτης Παύλα, εκπρόσωπος της Νότιας Όχθης της Μεσογείου, για να ε, σχολιάσει τις αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης, τις πρόσφατες. Δεν θα σχολιάσω λοιπόν αυτό το σκέλος, διότι δεν είναι ο δικός μου ρόλος και φαντάζομαι ότι εύκολα το αντιλαμβάνεστε. Θα ήθελα όμως να επανέλθω σε ένα θεμελιώδη ζήτημα. Χρειάζεται καθολική και ισορροπημένη προσέγγιση της μετανάστευσης. Δεν θα πρέπει να λησμονούμε όλη την εικόνα, την πραγματικότητα, ίσως είναι πολλοί λόγοι, δεν μπορώ να τους αναφέρω εδώ, αλλά είναι εκατομμύρια, εκατομμύρια εκείνοι που ζουν σήμερα στην Ευρώπη και κατάγονται από την νότια όχθη της Μεσογείου. Με τρόπο καθόλου ειρηνικό, νόμιμο και ενταγμένοι στις κοινωνίες μας. Και εδώ μιλώ για την συντριπτική πλειονότητα. Όταν μιλούμε λοιπόν για αυτές τις μετακινήσεις πληθυσμών θα πρέπει να το έχουμε υπόψη μας. Επίσης δεν λησμονώ τις πάμπολες εκθέσεις που δείχνουν ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση χρειάζεται εργατικά χέρια και τις επόμενες ε, δεκαετίες, δεκάδες εκατομμύρια. Είναι πάρα πολλέ οι εκθέσει και αναφέρουν και πολλά αριθμητικά στοιχεία. Επίσης δεν θέλω να λησμονήσω πόσο σημαντική είναι αυτή η ε, ανταλλαγή. Αν θέλουμε περιφερειακή συνεργασία, αυτή δεν είναι νοητή χωρίς ε, μετακινήσεις ε, πληθυσμών και πολιτών. Θα πρέπει λοιπόν να δούμε αυτό το θέμα της μετανάστευσης ενταγμένο σε ένα συνολικότερο ε, όραμα εξισορροπημένο έχοντας υπόψη τα εξή. Πρώτον, έχουμε ανάγκη να συνεργαζόμαστε. Δεν είναι λόγια το αέρα αυτά θεωρητικά. Επιτρέψτε μου να σας δείξω μια διαφάνεια που δεν πρόλαβα προηγουμένως. Εδώ. Αυτά είναι στατιστικά στοιχεία της Frontex που δείχνουν, βέβαια σταματούν στις αρχές του 2015, λείπει το πρώτο εξάμεινο του 2015, αλλά δείχνουν τους τρεις διαδρόμους. Υπάρχουν και άλλοι διαβλοί που έχουν στο μεταξύ δημιουργηθεί, βλέπε κεντρική Ευρώπη. Και βλέπουμε ποια προβλήματα ε, δημιουργήθηκαν πρόσφατα στα σερβο-ουγγρικά σύνορα. Λοιπόν υπάρχουν και άλλες ε, δύο... Ε, εδώ έχουμε λοιπόν το δυτικό διάδρομο που κυρίως αφορά το Μαρόκο και την Ισπανία όπου χάρη στη συνεργασία, χάρη στην εταιρική σχέση και χάρη σε μια πραγματική ε, κοινή προσπάθεια οι στατιστικές σήμερα δείχνουν ότι τα σύνορα ε, έχουν καλύτερη διαχείριση. Καλύτερη διαχείριση δεν σημαίνει έλλειψη προβλημάτων, αλλά σημαίνει ότι υπάρχουν δομές, κράτη, υποδομές. Και αν σήμερα υπάρχουν προβλήματα με ανθρώπινες τραγωδίες και δράματα στη Μεσόγειο, είναι επειδή υπάρχει το πρόβλημα που ονομάζεται Λιβύη. Γιατί εκεί δεν έχεις συνομιλητή. Σε ποιον αποταθείς για να αναπτύξεις ε, κάποιες συνεργασίες. Χρειάζεται λοιπόν η συνεργασία αυτή να είναι ε, δομημένη, διαρθρωμένη. Δεν είναι λόγια του αέρα όταν η ουσιαστική συνεργασία είναι και τα αποτελέσματα χειροπιαστά. Αλλά υπάρχει και ε, το θέμα της ανάπτυξης. Ο κόσμος γιατί μεταναστεύει. Για αντικειμενικούς λόγους που μπορεί να είναι πολιτική αστάθεια. Αλλά γιατί υπάρχει πολιτική αστάθεια. Το να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους. Και ε, όταν ονομάσουμε το πρόβλημα χρειάζεται και τη μετώπιση του. Στην ε, Αφρική, ας πούμε, νοτίως της Σαχάρας, όπου βλέπουμε να αυξάνονται οι μεταναστευτικές ροές, υπάρχουν δεδομένες πολιτικές καταστάσεις που χρειάζονται τη μετώπιση. Το ίδιο ισχύει και για τη μετανάστευση που ε, έχει οικονομικά κίνητρα. Αύριο θα έχουμε και κλιματικούς μετανάστες ε, θα πρέπει λοιπόν να έχουμε τη σύνολη εικόνα στο μυαλό μας για να προσπαθήσουμε να δώσουμε απαντήσεις. Να σας δώσω ένα συγκεκριμένο παράδειγμα από τη δική μας εργασία. Ε, το Ευρωμεσογειακό Πανεπιστήμιο στη ΦΕΖ του Μαρόκου απευθύνεται στους νέους, είναι περιφερειακή προσπάθεια, διασυνοριακή και απευθύνεται στους νέους για να γίνουν απασχολήσιμοι και αποδέκτες δεν είναι μόνο οι νέοι για να σταματήσει η λαθρομετανάστευση, αλλά για να ευνοηθεί και μια ποιοτική μετακίνηση που θα είναι αμοιβαία επωφελής. Προχωρούν τα έργα αυτά με ικανοποιητικό ρυθμό, αλλά θέλω στο μέλλον να αποτελέσει φάρο και εμβληματική προσπάθεια για να διευρυθεί ε, αυτό το έργο και να αποκτήσουμε ένα κοινό τρόπο σκέψης, μια κοινή κουλτούρα για να έχουμε πιο ποιοτική μετακίνηση, πιο ενάρετη ας πούμε. Επίσης, κάνετε ερωτήσεις για τις ελεύθερες συναλλαγές και τις επενδύσεις. Θα πρέπει να έχουμε εδώ διασταυρωμένα συμφέροντα. Τι σημαίνει αυτό. Στη Μεσόγειο δεν βλέπουμε μόνο προκλήσεις αλλά και ευκαιρίες και θα πρέπει αυτό να το αντιληφθούμε. Επιτρέψτε μου να το αναφέρω γιατί είναι το πιο πρόσφατο παράδειγμα όταν η Πεζό επενδύει στο Μαρόκο 600 εκατομμύρια ευρώ μόλις την περασμένη εβδομάδα. Αυτό δεν είναι αναπτυξιακή συνεργασία και μόνο, είναι εταιρική σχέση, αμοιβαία αμοιβαία-εποφελής και σημαίνει ανταγωνιστικότητα για την εταιρεία, την Peugeot, αλλά και τη διεθνή ανάπτυξη. Αυτά λοιπόν είναι τα κοινά διασταυρούμενα συμφέροντα και ε, μάλιστα αποτελούν την ισχύ αυτής της ε, γερής ε, περιφερειακής ολοκλήρωσης αμοιβαία εποφελούς, επαναλαμβάνω. Πολλά ερωτήματα έγιναν και ο χρόνος που μου δώσατε κύριε Πρόεδρε δεν μου επιτρέπει να απαντήσω σε όλα. Επιτρέψτε μου σύντομα σε δύο ε, ερωτήσεις συγκεκριμένα για την ευρωπαϊκή πολιτική γειτονίας. Θεωρώ συνάδελφοι ότι είναι μια πολύ σημαντική στιγμή. Πρέπει να κατανοήσουμε τη σημασία της πολιτικής γειτονίας η οποία να εδράζεται στην βάση της εταιρικής σχέσης. Έτσι, στα πλαίσια της έκθεσης για τη γειτονία, της ευρωπαϊκής πολιτικής για τη γειτονία, Διάβασα την έκθεση του κυρίου Κουκάν, τον συγχαίρω για το τι έχει κάνει μέχρι τώρα για τη γειτονία γενικότερα. Αλλά αν μπορώ μου επιτρέπετε να κάνω μια σύσταση είναι να ενισχύσουμε το περιφερειακό χαρακτηριστικό, την σημασία της περιφερειακής συνεργασίας έτσι ώστε να μην αυτοπεριοριστούμε σε μια γραμμική αντίληψη και η οποία μας περιορίζει στα διμερεί θέματα. Αλλά να συμπεριλάβουμε αυτές τις διμερείς δυναμικές σε ένα ευρύτερο γενικότερο στρατηγικό πλαίσιο. Έχει φτάσει η στιγμή η κατάλληλη γιατί οι προκλήσεις είναι περιφερειακές και περιφερειακές πρέπει να είναι και οι απαντήσεις. Τώρα για την πολιτική διάσταση τέθηκε το ερώτημα άλλωστε το θέμα της κοινοβουλευτικής συνέλευσης για την Ένωση της Μεσογείου. Η δυναμική αυτή πρέπει όχι απλά να διατηρηθεί αλλά να ενισχυθεί. Δεν θα πρέπει μόνο να ενισχύσουμε τις ε, ε, διαδραστικές αν θέλετε μορφές επικοινωνίας ανάμεσα στο Κοινοβούλιο το Ευρωπαϊκό και στην Ένωση και στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση όπως ακριβώς το είπα προηγουμένως και γι' αυτό εδώ η συνέλευση πρέπει να παίξει ένα ρόλο πολύ σημαντικό. Αν πρέπει κάτι να πω για να κλείσω και πέρα από τον κοινοβουλευτικό σοβινισμό εγώ είμαι περισσότερο ε, φανατικά υπέρ της Μεσογείου θα έλεγα περισσότερο από ποτέ όπως έλεγε και ο Μπεργαμινή προηγουμένως αυτό που έχουμε ανάγκη είναι μια δομή περιφερειακής συνεργασίας, μια δομή συνάντησης, από κοινού προσπάθειας. Τότε μόνο το μέλλον μας θα έχει τύχη. Αυτή η μέθοδος, αν θέλετε, συνεργασίας από κοινού προσπάθειας θα αποκτήσει νόημα. Αν δεν υπήρχε η Ένωση για τη Μεσόγειο θα έπρεπε άμεσα να τη δημιουργήσουμε. Ευχαριστώ τον Γενικό Γραμματέα. Ε, είμαστε για 8 χρόνια θα είμαστε μαζί. Θα συνεχίσουμε την προσπάθεια από κοινού. Σας ευχαριστώ πολύ. Και σας ευχαριστώ και για την παρουσίαση του προγράμματος δράσης της οργανώσεώς σας. Είστε επανειδήν.